Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που μπορώ να σας χαιρετήσω εδώ. Άρχισε η συνεδρίαση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πείσω στην προσοχή στο γεγονό ότι κατόπιν έχουμε ψηφοφορίε. Και βέβαια δεν θα χαρούν οι συνάδελφοι αν καθυστερήσουμε. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρονογόρευσης. Δεν θα είμαι πάρα πολύ ε, επίκης. Το πρόσημο σημείο της διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κάλλος Χωσέη Τούρκα Σανκούλου για εφαρμογή οδηγία για διαχείριση των αποβλήτων. Θα ήθελα αμέσω να δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να αρχίσω για αυτή την ε, έκθεση